ψηφίσουμε αύριο στις 12 το μεσημέρι την έκθεση αυτή. Και εδώ ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Η επόμενη θα διαξαρθεί Τετάρτη, αύριο, 12 Μαρτίου, στις 8.30, από τις 8.30 έως στις 2 και από τις 3 έως το, τις 11 το βράδυ. Η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα. Λίγη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ.